είναι η προφορική ερώτηση με συζήτηση, η πορεία προς τη δημιουργία Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Χαιρετίζω τον Επίτροπο Ταγιάννη και δίνω το λόγο στον κύριο Βιτάλ Μορέιρα, ο οποίος είναι ο συντάκτης της ερώτησης. Κύριε κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αυτή συνετάχθη πριν να ξέρουμε ότι θα αλλάξει η Επίτροπος Εμπορίου. Ελπίζουμε ότι ο νέος Επίτροπος θα απαντήσει το ερώτημά μου. Όπως ελέγχθη, η παρούσα ερώτηση αφορά το θέμα της δημιουργίας Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών έως το 2010. Στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελόνης αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το 2010 μία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στη Μεσόγειο και βασίζεται στο ότι υπάρχει η προσέγγιση που θα περιλαμβάνει το δίκτυο ελευθέρων συναλλαγών βορρά-νότου και ένα αντίστοιχο νότου-νότου. Είναι πολύ μακριά η πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Πιστεύει η Επιτροπή ότι η δημιουργία αυτή τη ζώνη ω το 2010 ήταν ρεαλιστικό στόχο. Εξ αρχή θα μπορούσε η Επιτροπή να μας αιτιολογήσει αυτή την απάντηση και να μας δώσει κάποια επιχειρήματα. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι πρόκειται σύντομα να εγκριθεί ένα νέο ευρωμεσογειακό χάρτη πορεία και ενδεχομένω ένα νέο μηχανισμό για να μπορέσει να διευκολυνθεί το εμπόριο και οι επενδύσει από την περιοχή. Μπορεί να μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε η Επιτροπή για τι ε, πραγματικέ πρακτικέ πτυχέ και τι συνέπειε τη εφαρμογή ενό τέτοιου μηχανισμού. Τρίτον, μπορεί η Επιτροπή να αναφερθεί στην πορεία της συμφωνίας του Αγαδίρ και να εξηγήσει με ποιο τρόπο προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει νέα πνοή σε αυτή τη συμφωνία και να ενισχύσει τη διάσταση νότου, νότου στα πλαίσια της δικασίας της Βαρκελόνης. Μπορεί η Επιτροπή επίσης να μας ενημερώσει με ποιο τρόπο ενσωμάτισε τις συστάσεις που είχαν γίνει Στη μελέτη που εκπώνησε το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις για την αηφορία και να λάβει υπόψη στις διαπραγματεύσεις την κοινωνική συνοχή και την αηφορονάπτυξη. Πέμπτο, μπορεί η Επιτροπή να μας εξηγήσει τι περιλαμβάνει η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία μετά το πάγωμα του 2004. Πέμπτο, μπορεί η Επιτροπή να μας πει τι ακριβώς γίνεται με τις διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη. Έβδομο. Κάποιες χώρες της Μεσογείου εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να διευρύνουν τις εμπορικές τους συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η Επιτροπή να μας ενημερώσει για τη νέα αυτή γενεά ε, συμφωνίων Δεύτερον, μπορεί να μα πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν στα πλαίσια των νέων ερευνητήτων τη ηθική της Λισαβόνα και στον τομέα αυτό του εμπορίου θα λάβει υπόψη ένα προηγούμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαπραγμάτευση, πριν από τη διαπραγμάτευση αυτών των νέων συμφωνιών. Αυτές είναι οι απαντήσεις που θα ήθελα να έχω στα ερωτήματά μου, κύριε Επίτροπε. Και δεδομένου ότι Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την διαδικασία της Βαρκελόνης και δεδομένης κατάστασης πιστεύω, σημερινής πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας έθεσα είναι πολύ επίκαιρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μωρέιρα. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριο Σταγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μωρέιρα απαντώ, σας απαντώ εξ ονόματος της Επιτρόπου Άστον. Όσον αφορά την ευρωμεσογειακή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μέχρι το 2010 βεβαίως είναι ρεαλιστικός στόχος και μέχρι τον επόμενο χρόνο θα δείτε ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έστω και αν πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η οικονομική ολοκλήρωση στην ευρωμεσογειακή ζώνη πρόοδοι έγιναν κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις Βορρά-Νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, με εξαίρεση την Συρία, έχει προχωρήσει σε διμερείς συμφωνίες σύνδεσης που αφορούν κυρίως ανταλλαγές αγαθών. Επίσης, πολυμερείς συμφωνίες όσον αφορά την προώθηση γεωργικών προϊόντων, ε, καθώς επίσης και για τον καθορισμό δεσμευτικών ε, διαδικασιών διαδικασιών για την λύση αντιπαραθέσεων. Περαιτέρω συμφωνίε θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2010. Όσον αφορά τις νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μεσογειακούς εταίρους, πρέπει να σας πω πάντα ε, στη διάσταση βορρά-νότου με την ευκαιρία ε, της συνεδρίασης ε, σε υπουργικό επίπεδο τη 10 η Νοεμβρίου έγινε συζήτηση για περαιτέρω ε, ανταλλαγή, ε, ε, περαιτέρω σχέσεις ανταλλαγής μέσα στα πλαίσια Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλογών που θα διευρυνθούν ακόμα περισσότερο μετά το 2010. Βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθούν και οι παρούσες διαδικασίες έτσι ώστε να αρθούν οι τεχνικές δυσκολίες ε, να λιανθούν προβλήματα τα οποία αφορούν, την, ε, ε, αφορούν θέματα υγειονομικά καθώς επίσης και θέματα αηφορίας και διαφάνειας το, Μαρόκο θα είναι ενδεχομένως ε, η πρώτη μεσογειακή χώρα με την οποία θα ξεκινήσει οι προγραμματεύσεις ήδη από τον επόμενο χρόνο και είναι προφανές ότι με την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενότατα με το Κοινοβούλιο ε, για θέματα εμπορίου. αλλά η Ευρωμεσογειακή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών έχει και μια διάσταση νότου-νότου. Δημιουργία δηλαδή ε, μία ζεσ μεταξύ των χωρών αυτών. Η διαδικασία του Αγαδίρ ξεκίνησε και αυτή είναι την συζήτηση γιατί, και αυτή τη διάσταση μάλλον για τις ευρωπαϊκές χώρες ε, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως το Ισραήλ ε, και την Τουρκία. Εκεί έχουν ξεκινήσει ήδη συμφωνίες ενώ για άλλες χώρες βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Είναι γεγονός πάντως ότι οι ανταλλαγές και οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων έχουν έχουν αυξηθεί έστω και αν δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο το οποίο επιθυμούσαμε και προβλέπαμε στην αρχή. Η έλλειψη ε, ε, τοπικής αγοράς ικανής ε, να προσελκύσει επενδυτές, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών θα, μετά το 2010 θα διευκολύνει διευκολύνει τις διαδικασίες. Επίσης ε, προβλέπονται και κάποιοι, πιο ε, μέσοπρόθεσμοι, βράχοι πρόθεσμοι μηχανισμοί. Ε, ας πούμε ο, ο μηχανισμός αυτός ο οποίος ε, θα δίνει έγκαιρα πληροφορίες όσον αφορά τους, της την ομοθεσία, όσον αφορά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, όσον αφορά οι ειδικέ συνθήκες που υπάρχουν στην Μεσογειακή ζώνη. Όσον αφορά τώρα την αηφορία στην οποία αναφερθεί αναφερθήκατε. Όπως ε, και σε όλες τις περιπτώσεις ε, ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια μελέτη ε, επιπτώσεων σχετικά με την αηφορία. Αυτή η μελέτη έλαβε χώρα το 2007 και χρησιμοποιείται και για τις παρούσες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και για τις μελλοντικές. Η ε, μελέτη αηφορίας λοιπόν όρισε κάποιες ε, περιόδους ε, οι οποίες αφορούν ειδικέ απαιτήσεις για, μεταβατική, για πρόβλεψη μεταβατικών περιόδων καθώς επίσης και για επιμήκυνση συμφωνιών που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Επίσης όσον αφορά την συζήτηση για την εγκατάσταση και για την παροχή υπηρεσιών κυρίως στη διάσταση συνεργασίας νότου-νότου και εκεί ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Όσον αφορά τη συμφωνία για την Συρία στην οποία έγινε λόγο. το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία αναθεώρηση τη συμφωνία Σύνδεσης έτσι ώστε να μελετήσει εάν πριν την τελική ολοκλήρωση της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης αυτής ε, χρειάζονται κάποιες τεχνικές ε, προσαρμογές. Ξεκίνησε λοιπόν συζήτηση με τους Συρίου συναδέλφου, έτσι ώστε να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα με τις νέες χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία ε, και ε, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και οι περαιτέρω συζητήσεις του 2004. Ε, η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 2008. Στην προηγούμενη εβδομάδα κοινοποιήθηκε η συμφωνία αυτή και είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την ε, Λιβύη, το Νοέμβριο του 2008 ξεκίνησαν ε, στις ε, Βρυξέλλες οι συζητήσεις για μια συμφωνία πλαίσιο για βάσει μιας, ενός φιλόδοξου προγράμματος ε, για την αρχή της εγκατάστασης, τη διευκόλυνση των υπηρεσιών ε, και η συμφωνία αυτή, ε, αυτή με την Λιβύη θα είναι το, η τελευταία ψηφίδα του μοσαϊκού. Διότι θα έχουμε πλέον με τη συμφωνία της Λιβύης θα έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική όσον αφορά την Ευρωμεσογειακή Ζώνη έστω και αν η Λιβύη δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως δε όσον αφορά το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο καθώς επίσης και τις υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει ειδικέ ε, συζητήσεις οι οποίες όμως βρίσκονται στην αρχή τους και θα χρειαστούμε χρόνο μέχρι ότου τις ολοκληρώσουμε. Σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Λιβύη για, την, για να μπορέσει να δημιουργήσει τις υποδομές αυτές οι οποίες θα τις επιτρέψουν να γίνει εμπορικός εταίρος στο ίδιο επίπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταγιάννη. Και προχωράμε τώρα στους ομιλητές εξονόματος πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Παπαστάμκος. Τον, ε, την στρατηγική σημασία ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση για την εμπέδωση της πολιτικής, της οικονομικής και της πολιτισμικής συνεργασίας και γενικότερα της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ε, περιοχή. Καλούμε τους Υπουργούς να υιοθετήσουν στην προσεχή διάσκεψη οδικό χάρτη για την πραγμάτωση της Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Η διμερής προσέγγιση πρέπει να συνοδευτεί από μια περιφερειακή προσέγγιση. Επίσης, πέραν της διάστασης βορρά νότου ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ την οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση νότου νότου στην οποία αναφέρθηκε τόσο ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου ο κ. μορέιρα όσο και ο επίτροπος ο κ. σταγιάννη. τονίζω ιδιαίτερα την ανάγκη ενσωμάτωσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών προνοιών και φυτοϊγειονομικών προτύπων που θα πρέπει να συνοδεύουν το άνοιγμα των αγορών. επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα που αφορούν στι εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά τάσσομαι υπέρ τη ενίσχυση τη διαδικασία τη Βαρκελόνη και Ένωση για τη Μεσόγειο, καθώ και των προγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί εντό του πλαισίου τη σε στρατηγικού τομεί, όπω είναι η συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Τέλος, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των θαλασσίων διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση που είχε υποβάλει η Ελλάς το περασμένο καλοκαίρι για την εγκαθίδρυση ενός παρατηρητηρίου μεταφορών στην ε, Ανατολική, Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αρίφ Καντάρ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βιτάλ Μορέιρα για την παρέμβασή του στις 9 ε, Δεκεμβρίου θα συζητήσουν οι Υπουργοί Πορείου το θέμα της αναθέρμανσης των εμπορικών μας Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνουμε την εξής ε, διαπίστωση. Εάν έπρεπε η δημιουργία αυτής της ζώνης ελευθέρου εμπορίου και ελευθέρων συλλαγών να είναι υποφελής για όλους, θα είχαμε κάνει κάτι διαφορετικά, διότι βλέπουμε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν θα συμβεί το ίδιο για αυτούς που είναι στην βόρεια ή στην νότια πλευρά της Μεσογείου. Θα ήθελα να Υπενθυμίζω τους τρεις πυλώνες, τον πολιτικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό και θα έπρεπε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον ε, οικονομικό και εμπορικό τομέα να παραγνωρίσουμε κάπως την πολιτική σημασία. Πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, σταθερότητα όμως και ειρήνη. Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Δεν το πιστεύω διότι και τα ίδια τα γεγονότα μιλούν για αυτή την πραγματικότητα. Η η δημιουργία ευρωμεσογειακής ζώνης θα είχε ως στόχο να κάνει αναθέρμανση της κατάστασης η οποία περνάει από μια στασιμότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι η πολιτική μας κάνει να έχουμε ελπίδες. Είμαι υπέρ αυτών που είναι υπέρ της διαδικασίας της Βαρκελόνης και αυτών που πιστεύουν ότι η πρόοδος δεν μετράται μόνο με τις στρατιστικές. Το εμπόριο για το εμπόριο, όχι, δεν το πιστεύω. Το εμπόριο όμως ε, για να εξυπηρετηθεί η, η οικονομική ανάπτυξη, η ευημερία όλων ε, και είναι κάτι το οποίο πιστεύω, αλλά θα πρέπει οι διαπραγματεύσει να στραφούν προ αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό στην επόμενη συνάντησή σα θα ήθελα να σα πω να είστε συλλογικά υπεύθυνοι, να μην αρκεστείτε μόνο σε τεχνικού περιεχομένου συζητήσει για την άρση των εμπορίων στο εμπόδιο. Δεν θα πρέπει μια τέτοια κατάσταση να διενιστεί. Σήμερα πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσει στην οικονομική κρίση, στην απώλεια θέσεων απασχόληση και να προσέξουμε την ανάπτυξη τους ε, προστασίες του περιβάλλοντος και να γίνουν όλες οι πολιτικές μας ανθρωποκεντρικές. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρινάλντι, ένα λεπτό. Ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω με μία φράση από τις χίλιες και μια νύχτες δεν υπάρχει στασιμότητα για αυτόν που ε, λέει λοιπόν δεν υπάρχει στασιμότητα. Ε, αυτός ε, που, που μένει σταθερός δεν είναι πραγματικός. Οπωσδήποτε πρέπει να κινείται. Κινείται οποιοδήποτε θέλει να απομακρυνθεί από την φθορά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θυμηθούμε λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την ευρωμεσογειακή ζώνη συνεργασίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα σε Αυτή τη στιγμή το 50% του πληθυσμού της ε, Νότιας ε, Μεσογείου ε, έχουν ηλικία κάτω των 20 ετών. Και επίσης ότι αναφερόμαστε σε ένα δις ε, ε, ε, πολιτών. Επίσης εμείς θέλουμε σαν φίλε ελεύθεροι να δώσουμε στους πολίτες αυτών των χωρών συνεργασίες οι οποίες δεν θα είναι γραφειοκρατικές και οι οποίες όμως δεν θα δίνουν χρήματα στις ολιγαρχικές, στα ολιγαρχικά καθεστώτα τα οποία πολύ συχνά βρίσκουμε επικεφαλής αυτών των χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από κάποια χρόνια διαπραγματεύσεων στη διαδικασία τη Βαρκελόνη, έχουμε σοβαρέ αμφιβολίε του γεγονό ότι η διαπραγμάτευση μια συμφωνία ελευθερωση συναγών τύπου Euromed είναι η απάντηση στα προβλήματα τα οικονομικά, τα πολιτικά και τα προβλήματα ανάπτυξη περιοχή. Η μελέτη σκοπιμότητα απέδειξε ότι υπήρχαν δυνητικά πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες αρνητικών επιπτώσεων ε, στον κοινωνικό, στον περιβαλλοντολικό και στον τομέα της ε, περιφερειακής ένταξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύουμε πραγματικά ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον οδικό χάρτη του 2010 και μετά είναι πραγματικά μονοσήμαντη και δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο συζητείται σήμερα κυρίως διότι θέτει όλα αυτά τα θέματα των κοινωνικών επιπτώσεων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην ε, περιφερική άντεξη. Διότι στην παράγραφο 10 ζητά αναθεώρηση των ε, εμπορικών συμφωνιών και της κοινωνικής πτυχής και της περιβαλλοντικής πτυχής πιστεύουμε ότι αν αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτή την εμπορική συμφωνία που θέλουμε να επιτύχουμε στην διαδικασία της Βαρκελόνης. Ευχαριστώ ο κύριος Μέιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την ομάδα μου είναι αδύνατον το εμπορικό μέρος να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε από την πολιτική διάσταση, από τη διάσταση του προβλήματος που αφορά μετανάστες. Γι' αυτό είμαστε κατά του να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση και με το Μαρόκο και με το Ισραήλ. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο πιο απαιτητική για την προάσπιση των αξιών που θα μας οδηγήσουν σε μοιρασμένη ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή στο Λανθαρότε κάνει απεργία πίνεις μία πολίτη από το Σαχαράουι, διότι έχει προβλήματα με το Μαρόκο. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και απαιτεί από τα κοινοτικά όργανα μία σοβαρή στάση κατά του βασιλιά του Μαρόκου. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει μόνο να κοιτούμε τα συμφέροντα του εμπορίου, αλλά ενδιαφερόμαστε κυρίως για την πράξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά ο κόμις του Ντάρτμουθ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κόμμα της ανεξαρτησίας της Ευρώπης είναι κατά της συμφωνίας ε, της Ευρωμεσογειακής διότι θα προσφέρει σημαντικές εμπορικές υποχωρήσεις και επιδοτήσεις σε μη κράτη-μέλη. Και αυτό οπωσδήποτε θα είναι σε βάρος άμεσο ή έμεσο του Ευρωπαίου Φορολογουμένου. Επίσης, όταν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μίλησε στην, Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου, στην Επιτροπή Εμπορίου ε, για την Ευρωμεσογειακή είπε και παραθέτω αναμφίβολα δεν τίθεται θέμα εφαρμογής όλων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέχισε και είπε ότι η εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι επιλεκτική και ευφυής. Σε αντίθεση εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεχτήκαμε και μάλιστα υποφέρει η οικονομία μας από αυτό, δεχτήκαμε την εφαρμογή όλων των κοινοτικών κανονισμών και μάλιστα σε εμά εφαρμόζονται με τρόπο μη ευφυή και καθολικό. Ούτε καν μας επετράπει να έχουμε τις κλίδες ασφαλείας που θα θέλαμε. Ε, αλλά δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Μετά τη Λισαβόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο εμείς θα... Ε, ε, ε, ε, υποφέρομαι ε, μετά από την ε, κάλυψη των υψηλών αξιωμάτων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της ΥΠΑ του εκπροσώπου, η οποία ήταν ε, στο CND ε, η εκπρόσωπος των πλέον αριστερών απόψεων. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα μας εκπροσωπήσουν. Οι ευρωμεσογειακές χώρες όμως δεν θα αντιμετωπίσουν ε, τα, τη ζημία από την πολιτική αυτών των υψηλών προσώπων. Ε, ας δούμε τις χώρες για τις οποίες συζητούμε, η Συρία και η Λιβύα από όλες τις χώρες ε, ε δέχτηκαν εμπορικές υποχωρήσεις και ε, επιδοτήσεις. Ε, τι διασφαλίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν, πουθενά. Και οι δύο χώρες έχουν ε, μακρά και πραγματικά επονίδιστη πορεία και ιστορία. Αυτό το τμήμα ε, του ψηφίσματος ε, ε, κατεγράφει πραγματικά μέσα σε μία παραζάλη και γι' αυτό εμείς τα σώμεθα κατά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπονσινιόρ δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Γιώργ Λάιχτφιλντε για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ελεύθερο εμπόριο, οι ελεύθερες συναλλαγές είναι καλές ε, αν δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτό το θέμα. Πρόκειται για κάτι παραπάνω εδώ. Δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Θα πρέπει να φροντίσουμε για βιώσιμες αηφόρους επιπτώσεις. Θέλουμε ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να δημιουργηθεί ευημερία για όλους μέσα από αυτή την πολιτική. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικότερο από το να φροντίσουμε ε, μόνο την απελευθέρωση των αγορών, το άνοιγμα των αγορών ε, από το οποίο ίσως λίγοι μόνο θα ωφεληθούν. Αν θέλουμε να απελευθερώσουμε το εμπόριο, ο στόχος ε, της προσπάθειας και σε εμά και στου νότιου γείτονε, ο στόχο θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση τη ανεργία. Κυρίω όταν ε, οι γυναίκε, οι νέοι, ε, ο πληθυσμό τη υπαίθρου θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερε ευκαιρίε. Αν αυτό είναι ο στόχο μα, τότε θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αν ο στόχο μα είναι αποκλειστικά η απελευθέρωση, το άνοιγμα των αγορών και η αποκόμιση κερδών μόνο από ορισμένου, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, την, για τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Μπονσινιόρε, από ό,τι με ενημερώ... Α, ο κύριος Σικέρσκι θα μιλήσει για 1,5 λεπτό και για τον κύριο Μονσινιόρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος στόχος της συμφωνίας Euromed είναι να υπάρχει πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών της Μεσογείου και να ενισχυθεί η οικονομία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει και τις αραβικές χώρες ώστε να μπορέσει να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της Βαρκελόνης και να λάβουμε υπόψη και το κράτος δικαίου και την δημοκρατία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνιών των κρατών αυτών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου, η απελευθέρωση του εμπορίου με την παροχή αγροτικών προϊόντων από τις χώρες αυτές θα ενισχύσει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις εξαγωγές σιτηρών, φρούτων, λαχανικών και κρέατος στην περιοχή. Η μεσογειακή συνεργασία χρειάζεται πολλές προσπάθειες εκ μέρους όλων των ε, συμμετεχουσών χωρών. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Catch the ο κύριος Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από κάποιες εβδομάδες ήμουν σε μια συνεδρίση μια καναδική αντιπροσωπεία που συζητούσε ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγουμένω κάτι τέτοιο συζητήθηκε για την Νότια Κορέα. Σήμερα συζητούμε κάτι που παρεμφεραίνει το Euromed. Μπορεί η Επιτροπή να μα πει πόσου τέτοιου είδου συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, πού είναι τα κέρδη από τη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, Ποιες είναι οι ευκαιρίες που δίδονται για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες από την πλευρά της οικονομική και από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και ίσως δεν συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν, αλλά το κύριο αλλά θα ήθελα σε θεμελιώδη σημασία θέματα και αφήνοντας κατά μέρου κάποια δευτερεύοντα να μας δώσετε απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κυρία Ντότ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου. Βρίσκομαι ενώπιον σας απόψε ως μια Ευρωπαία που πιστεύει στη συνεργασία των εθνών. Όχι ε, ως Ευρωπαία που πιστεύει στο φεντεραλισμό του προγράμματος αυτού για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Λισαβόνα, θα μειώσει τη δυνατότητα που έχουμε να διεξάγουμε εμπόριο με όποιον θεωρούμε σκόπιμο. Επίσης, ε, συρρυκνώνεται η δημοκρατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συσχετίζεται με τις, περασμένες, τις εξελίξεις της ε, περασμένης εβδομάδας ε, την ε, ε, εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Υπουργού, της Υπουργού των Εξωτερικών. Αυτή δεν είναι ε, μια κατάσταση η οποία υποθέτω θα βρίσκει σύμφωνη την Κομισιόν και με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις απόψεις της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεραίρο. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την θέσπιση ε, της Ευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Μία γενική που αφορά τις νότιες και ανατολικές χώρες της Μεσογείου και τις αναπτυσσόμενες χώρες που θέλει να αναπτύξει σχέσεις η και με τις χώρες ΑΚΕ. Ο Λακορντέρ από τη... είπε το εξή. Μεταξύ ισχυρού και αδύναμου, μεταξύ πλούσιου και φτωχού, η ελευθερία μπορεί να, η φτώχεια μπορεί να είναι σκλαβιά και ο πλούτο ελευθερία. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Στην απελευθέρωση του εμπορίου ιδίω σε ευαίσθητου τομεί όπως η Ελία και η Εργοστία είναι κάτι το οποίο έχει ε, δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην παρούσα οικονομική κρίση, διότι δημιουργεί προβλήματα στου πιο φτωχού για τα κοινωνικά δικαιώματα, για την απασχόληση και δημιουργεί προβλήματα σε θέματα επισητισμού. Για να ε, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε ώστε να υπάρχει καλή άποψη για όλου. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Παλαιστίνη και στην Ανατολική Σάχαρα που δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε στα πλαίσια τη συζήτηση που κάνουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα να λάβει κάποιος ξανά το λόγο. Παρακαλώ μου στηρίστε κύριε, ο κύριος Λάιχτφελ και ο κύριος Άριφ θα λάβουν το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συντομότερος από ένα λεπτό. Μία ερώτηση στον Επίτροπο. Συμφωνούμε ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν περιορίζονται στο εμπόριο. Έχουν άλλους στόχους ή και άλλους που μας βοηθούν όλους. Ρωτώ λοιπόν σε ποιο βαθμό η διαδικασία αυτή οδηγεί σε ε, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα, καλύτερη κατανομή του πλούτου. Μπορούμε, έχουμε κάποιες ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση και πόσο χρόνο θα ε, διαρκέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ο κύριος Σαρίφ. Θα ήθελα να πω κάτι στην κυρία Ντότς, να διαβάσει η συνθήκη της Λισαβόνας, διότι αν υπάρχει μια επιτροπή που θα ενισχυθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερη σημασία του επόμενου μήνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριο Μωραήρο έθεσε στον Επίτροπο μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και είπε ο κύριο Ταγιάννη, η Λιβύη και η Συρία ε, είναι χώρες για τις οποίες δεν δόθηκε απάντηση. Ε, εκεί όμως το θέμα της πρόσφυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό. Σας παρακαλούμε λοιπόν να απαντάτε σε τέτοιου είδους ερωτήματα που αφορούν την ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, το να μιλάει κανείς για την Ευρω... Μεσογειακή Ζώνη ε, ελευθέρου πορείου χωρίς ε, να αναφέρει το θέμα του προβλήματο μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ ε, δεν είναι σωστό. Θα ήθελα και γι' αυτό να μου μιλήσετε εδώ μέσω βαρύτητας του προβλήματος αυτού στην περιοχή να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος του Catch Θα δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτές, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επίτροπος Άστον απουσιάζει όχι λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει από τις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά γιατί είχε άλλες θεσμικές δεσμεύσει ε, λόγω της αντιπροεδρίας και του φακέλου με τον οποίο ασχολείται τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις περιπτώσεις που δεν θα μπορέσω να απαντήσω θα σας σταλούν οι απαντήσεις γραπτά. Ε, θα σταλούν λοιπόν προς όλους τους βουλευτές και θα τις έχουν στείλει η κυρία Άστον και οι υπηρεσίες της. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια δέσμευση η οποία αποτέλεσε πάντα επίκεντρο κάθε, κάθε δράσης κυρίως ε, όσον ε, αφορά ε, διαπραγματεύσεις με την Αφρική. Πάντοτε λοιπόν θελήσαμε η προτεραιότητά μας να αφορά την εγγύηση της πολιτικής σταθερότητος, ε, ο σεβασμό, τον σεβασμό των κανόνων και βεβαίως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία της δέσμευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολουθούν ε, βεβαίως όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν το εμπόριο, τις εμπορικές συμφωνίες, οικονομικές συμφωνίες. Επομένως, να καθησυχάσω τους βουλευτές ότι ουδέποτε και ουδόλως υποτιμάται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις όποιες συμφωνίες ή συζητήσεις ε, γίνονται με χώρες ε, με ε, έχουμε διαπραγματεύσεις και βεβαίως κάνουμε πάντα ε, και ελέγχους ε, και ε, συνεχίζουμε τους ελέγχους και ακόμα και μετά τις συμφωνίες. Όσον αφορά την Συρία, η Συμφωνία Σύνδεσης σε γενικές γραμμές ακολουθεί την μορφή άλλων συμφωνιών σύνδεσης της Ευρωμεσογειακής Ζώνης. Προβλέπει δηλαδή διάλογο σε κοινωνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε τακτικά διαστήματα Επίσης, προβλέπει δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών σε 12 το πολύ χρόνια, καθώς επίσης ε, ε, περιέχει και μακρόπνοες, μακρόπνοα προγράμματα σε πολλούς τομείς ε, καθώς ε, επίσης και στο θέμα ε, των, και σε θέματα τα οποία δεν αναφέρονται σε άλλες περιπτώσεις ιδιαίτερα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα διαγωνισμούς και προμήθειες εμπορικές συμφωνίες φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, γαλακτοκομικά μετά από μια σειρά ετών δύσκολης συνεργασίας και σχέσης με την διεθνή κοινότητα, η Συρία έκανε πολύ σημαντικά βήματα έτσι ώστε να προσεγγίσει τους ξένους εταίρους. Ε, και σαν υπουργό Μεταφορών ε, πήγα πρόσφατα και στην Λιβύη και διαπίστωσα ότι πραγματικά υπάρχει μια αλλαγή κλίματος Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την ε, Λιβύη, οι Λίβοι δέχονται ε, την αρχή και το περιεχόμενο των νομικών κειμένων όσον αφορά την ανταλλαγή αγαθών, ε, καθώς επίσης και εμπορικές συμφωνίες και κανόνες που αφορούν τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς, έτσι όπως αναφέρονται εις το κοινοτικό και κτημένο. Αλλά βεβαίως, όπως είπα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαγρύπνει πάντοτε. Ε, δεν ξέρω εάν απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας όσον αφορά τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό ε, συν ε, συζητήσεων για δημιουργία ζωνών ελεύθερων συναλλαγών. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θα έχετε σαφέστερες και πληρέστερες απαντήσεις μέσω γραπτού κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ταγιάννη. Ενημερωτικά σας πληροφορώ ότι λάβαμε πέντε ψηφίσματα επί του θέματος. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση σε αυτό το σημείο και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Επιτρέψτε μου να περάσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης προφορική ερώτηση για την ασφάλεια και διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος. Δίδω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπράιαν Σίμψον, τον συντάκτη της ερώτησης, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.